Τώρα, περνάμε στην ψηφοφορία. Πρώτο ψήφισμα αφορά το σχέδιο νόμου της Καμπότζης για τις ΜΚΠΑΟ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα ψηφίσουμε επί όλου του κειμένου του ψηφίσματος αυτού. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο ψήφισμα. Για την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και ιδιαίτερα υποθέσει, περιπτώσει Ιβ Μακβαμπάλα, Φρεντ Μπάουμα. Έχουμε το κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε, ελπίζω, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα, το κοινό ψήφισμα. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα για την περίπτωση των Απλερατζάπ, τον Μπαχρέιν. Μετά την ετολική σκέψη έχουμε τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε Α, θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Mm. Απορρίπτεται η τροπολογία 1 με ισοψηφία. Περνάμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία στο σύνολο του πρώτης ψηφίσματος. Να ψηφίσουμε, Ψήσατε όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε λοιπόν τώρα. Głosowania e, dotyczącego Sudanu, sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów. Περνάμε λοιπόν στο ψήφισμα για την κατάσταση δύο χριστιανών ιερών στο Σουδάν. Μετά την παράγραφο 3 στο κοινό ψήφισμα έχουμε την τροπολογία 3 από το ΕΛΚ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Μήπως καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 7, αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 αρχικό κείμενο. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Από την κυρία Βερζιά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Χτες το βράδυ έμαθα ότι τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης στο Σουδάν του κόμματος του Κογκρέσου καταδικάστηκαν σε 20 ραπισμούς τη Δευτέρα. Αμέσως εκτελέστηκε η ποινή έξω από το δικαστήριο. Στη χώρα αυτή νομίζω είναι ιδιαίτερη ταπείνωση αυτό και ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει και αυτό το νέο γεγονός στο ψήφισμα και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, είναι συνεργατικό αυτό. Θέλει κάποιος ε, να φέρει αντιρρήσει αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω κάποιον να, να διαφωνεί. Επομένω, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της τη παραγράφου 8, όπως ε, τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Στην αιτιολογική σκέψη 9, αιτιολογική αναφορά 9 μάλλον, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη F έχουμε τροπολογία 1 του ΕΛΚ ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 του ΕΛΚ ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το, την σκέψη H αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία η οποία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα αυτό με τεράστια πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης